Ε, ρυθμιστικό όφελος ε, που μπορεί να έχει σε μεγαλύτερο βαθμό ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, από τον φόρο δραστηριοτήτων, τον FAT. Τα δύο ερωτήματα θέλω να σας κάνω. Το πρώτο σε ό,τι αφορά το διαφορετικό tax rate. Είπατε και στα slides που μας δείξατε, κάνατε λόγο ε, για ένα rate της τάξης του 0,1% σε ό,τι αφορά τα ομόλογα και τις μετοχές και 0,01% σε ό,τι αφορά στα παράγωγα. Σε συνδυασμό βεβαίως και με τις νέες ρυθμίσεις για την αγορά παραγόγων γιατί στόχος ακριβώς ε, δεν είναι ε, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ενός τέτοιου φόρου κυρίως είναι να συμβάλλει ένας τέτοιος φόρος στην καλύτερη ρύθμιση προϊόντων και συναλλαγών που μέχρι σήμερα δεν ήταν επαρκώς ρυθμισμένα. Θα περίμενα, ε, θέλω να σας ρωτήσω, θα περίμενα ε, το αντίστροφο εφόσον θέλουμε να αποθαρρύνουμε συναλλαγές υψηλή ε, υψηλής συχνότητας, ίσως το rate για τα παράγωγα να έπρεπε να είναι μεγαλύτερο παρά τη συχνότητα από ότι για τα ομόλογα και τις μετοχές αυτό ήθελα να σας ζητήσω αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε. το δεύτερο εάν ε, βλέπετε κάποιες εξαιρέσεις αν θεωρείτε ότι κάποια, ε, κάποιες, κάποιοι τύποι συναλλαγών okay, κάποιοι τύποι συναλλαγών μπορούν ε, και πρέπει να εξαιρεθούν και το τρίτο και κλείνω γιατί πιστεύετε ότι μακροπρόθεσμα θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις από έναν ευρωπαϊκό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αυτό που μας παρουσιάζεται είναι καλά νέα. Χρησιμοποίησατε κάποια επιχειρήματα. Είχαν ακουστεί και ακουγόταν επί πολύ χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπερασπίστηκε η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, τι μπορούμε να πούμε, σας υποστηρίζουμε προφανώς. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε αυτή την απάντηση. Πρέπει να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια δεδομένη τη κρίση. Είναι μια απάντηση που επιθυμεί εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντω υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα έχουμε κάποιε επικρίσει, έχουμε να σα ζητήσουμε διευκρινήσει και θέλουμε να ζητήσουμε και την άποψή σα για ορισμένα θέματα φυσικά. Η συζήτηση δηλαδή δεν έχει γίνει. Ήδη το ερώτημα που ακούστηκε τους συντελεστές, τους φορολογικούς συντελεστές και την ελαστικότητα. Γιατί διαλέξατε αυτούς τους συντελεστέ. Θέλω να επανέλθω επίση στο θέμα της νομικής βάσης. Διαλέγετε τους ίδιου σπόρους. Πιστικό είναι, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητε. Όταν γίνουν οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, θα δείτε ότι πρέπει να τα πείσετε τα κράτη-μέλη και εμεί θα προσπαθήσουμε να σα βοηθήσουμε για να τα πείσετε. Θα πρέπει να τα πείσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συγκεκριμένη φορολογική βάση. Υπάρχουν μια σειρά από νομοθετικέ δυνατότητε και φορολογικέ δυνατότητε που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και που αποτελούν διαφορετικέ εναλλακτική λύση. Αλλά ο φόρος ε, που θα ενταχθεί στους ίδιου πόρου είναι μια καλή ιδέα. Έπειτα, τι χρονοδιάγραμμα σκέφτεστε για την εφαρμογή αυτού του μέτρου γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όσο πιο γρήγορα αποφασίσουμε, τόσο καλύτερα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τόσο καλύτερα θα είμαστε εξοπλισμένοι να καταπολεμήσουμε την κρίση και να μοιραστούμε πιο δίκαια το άχθος λόγω της κρίσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν είδα την παρουσίασή σας, κύριε Επίτροπε, ε, είπα, η πρώτη μου αντίδραση ήταν θα τον μηνύσω, γιατί μου έκλεψε τις ιδέες. Ε, τελικά όμω ε, δεν είναι πράσινο κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα το κάνω. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν. τέλο πάντων, α περάσουμε στα σοβαρά τώρα. Πέρα από το θέμα των συντελεστών, που συμφωνώ με την Άννη και τον Ούντο, αυτό που αμφισβητώ είναι μία από τις δηλώσεις που γίνεται στις διαφάνειές σας, που λέτε ότι η επίπτωση ε, στο ΑΕΠ, όπως κάθε φόρου, είναι αρνητική. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος βέβαια, αλλά οι άλλοι ευρωβουλευτές είναι. Είναι η πρώτη φορά που ακούω κάτι τέτοιο ότι υπάρχει συσχετισμό μεταξύ του επίπεδου φορολογίας και της ανάπτυξης του ΑΕΠ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θετική ή αρνητική σχέση ανάμεσα στα δύο. Τούτου λεχθέντος μπορούμε να πούμε ότι ποτέ δεν αρκεί κάτι. Αν καταφέρετε όμως να δρομολογήσετε αυτή την πρόταση, μπράβο σας. Πέρα από τα δύο πράγματα τώρα που ανέφερα, η αρνητικη σχεση αναμεσα στα δυο τουτου λεχθεντο μπορουμε να πουμε οτι ποτε δεν αρκει κατι αν καταφερετε ομως να δρομολογησετε αυτη την προταση μπραβο σας περα απο τα δυο πραγματα που ανεφερα η πραγματικη μου ερώτηση είναι εξή. Ε, θέλω να χαιρετήσω τους θαραλέου δεξιούς ε, προβουλευτές που αποφάσισαν να έρθουν σε αυτή τη συζήτηση. Σοβαρά το λέω. Υπάρχουν λίγοι από εσά και αυτό είναι ενδεικτικό. Τουλάχιστον εσεί είχατε το φέρος να έρθετε. Τώρα είναι η ώρα ε, να δείξετε και να πείτε τις απόψεις για την οικονομική διακυβέρνηση και ότι δεν θέλετε μόνο λιτότητα. Όταν λέτε ότι θέλετε ισορροπημένου ε, προπολογισμού. Θέλετε, αυτό σημαίνει ότι θέλετε και περικοπέ στον προπολογισμό, αλλά ότι θέλετε να προβλέψουμε και του κατάλληλου πόρου. Δεν είναι κανένα από του φιλελεύθερου όμω. Αυτοί όλο για την οικονομική διακυβέρνηση κραυγάζουν. Αλλά δεν είναι κανεί εδώ παρόν. Κανεί δεν έρχεται εδώ να μιλήσει υπέρ τη εξισορρόπηση των προπολογισμών. Ήρθε η ώρα τη αλήθεια τώρα. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώ θα αντιδράσουν όλοι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ευχαριστώ. You have the floor. Okay. Uh, uh, well, so I, I, I will, I will answer those uh, first questions. Ας απαντήσω αυτές τις πρώτες ερωτήσεις για τους φορολογικούς συντελεστές. Όταν μιλάμε για παράγωγα, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μετεγκατάστασης, αν οι συντελεστές είναι πολύ ψηλοί. Όταν μιλάμε δηλαδή, για αυτό το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο αν επιβληθεί μόνο στην Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος μετεγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους συντελεστές ως ενδεικτικούς δεν είναι απόλυτοι οι συντελεστέ αυτοί. Φυσικά θα του δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε την νομοθετική πρόταση. Υπάρχει δυνατότητα, Φερρυπίν, να έχουμε διαφοροποιημένους συντελεστέ. Για παράγωγα που τα διαπραγματευόμαστε στη ρυθμισμένη αγορά ή παράγωγα ή προϊόντα που τα διαπραγματευόμαστε εκτός ρυθμισμένης αγοράς. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. από την προοπτική των χρηματαγορών. Δεν είναι δεδομένοι και τελεσίδικοι αυτοί οι φόροι, αυτοί οι φορολογικοί συντελεστέ. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Πάντως είναι ελάχιστοι οι συντελεστές αυτοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ απαντάω μερικέ στο ερώτημα του κ. Μπούλμαν για τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έσοδα των εθνικών προϋπολογισμών. Πρόκειται για ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές και τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να πάνε στους ίδιους πόρους ενώ θα μπορούσαμε να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να θέσουν υψηλότερους ε, φορολογικούς συντελεστές από αυτούς τους ελάχιστους και τη διαφορά να τη χρησιμοποιήσουν για τους εθνικούς προπολογισμού. Να πάει δηλαδή στους εθνικούς προπολογισμού. Είναι σημαντικό και τα κρατημέλη εξάλλου. Όταν εισαγάγουμε ένα τέτοιο φόρο, στα πλαίσια των ιδίων πόρων, αυτό σημαίνει ότι και η συνεισφορά των Ακαθάριστον εγχώριων προϊόντων θα μειωθεί. Και επομένως αυτό θα είναι και θετικό για τη μείωση των ελλημάτων τους. Νομίζω ότι είναι και προ όφελο λοιπόν των κρατών μελών να έχουν θετική στάση απέναντι σε αυτό το φόρο. Και απέναντι σε αυτήν την πρόταση γενικά. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με τις υπηρεσίες μας επί της νομοθετικής πρότασης. Αυτό σημαίνει ότι θα υποβάλουμε ένα σχέδιο οδηγίας για το φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών το φθινόπωρο του 2011. Αυτός είναι ο στόχος μας. Φυσικά δεν μπορώ να δεσμευτώ τώρα, γιατί θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στο Σώμα των Επιτρόπων. Αλλά αυτή είναι η ιδέα καταρχήν. Να παρουσιάσουμε την πρόταση το φθινόπωρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις. Ανέφερα ήδη ότι προσπαθούμε να σχεδιάσουμε το φόρο με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να υπάρχουν αντισταθμίσματα. Δηλαδή, οι μη χρηματοπιστωτικές οντότητες ή οι πολίτες μπορούν να εξαιρούνται από αυτόν τον φόρο. Φυσικά θα υπάρχουν συναλλαγές που τις κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή άλλα όργανα. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα προτεθούν και εξαιρέσει. Αλλά δεν θέλω τώρα να επεκταθώ περαιτέρω για όσο αφορά το εύρο των εξαιρέσεων. Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλήσουμε για εξαιρέσει, για να μην δημιουργήσουμε καταστάσει που θα επιτρέψουν να μεταφερθεί ο φόρο. Δηλαδή από τα φορολογητέα πρόσωπα στα μη φορολογητέα πρόσωπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν σχεδιάζεται ένας φόρος. Για την επίπτωση τώρα του φόρου στο ΑΕΠ, όταν σας παρουσίασα την πρόταση, ε, εννοούσα ότι αν εξετάσουμε χώρια τον φόρο αυτό, μεμονωμένα, μπορούμε να συνάγουμε αυτό το συμπέρασμα ότι έχει αρνητική επίπτωση στο προπολογισμό. Υπάρχουν φυσικά διαφορετικοί τρόποι να τον αναλύσουμε, να τον εξετάσουμε. Δηλαδή, εξετάζουμε τα έσοδα από όλου του φόρου και κυκλοφορήσουμε σαν στην οικονομία, τότε μπορεί ε, η επίπτωση της κυκλοφορίας αυτών των φόρων να είναι συνολικά θετική. Αλλά αν κοιτάξουμε μεμονωμένα τον κάθε φόρο, σίγουρα το αποτέλεσμα είναι αρνητικό επί του, επί του ΑΕΠ. Euh, θα ξεκινήσω με... θα συνεχίσω μάλλον με τους εγγεγραμμένους του ΕΛΚΑ. Παλώνε. Τάισεν, Χουντής. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Πάντα ακούμε μεγάλη προσοχή τον κύριο Λάμπερτ όταν μιλάει και εγώ δεν αισθάνομαι δεξιό. <laughs> το λέω, ευθύ εξ αρχής. Απλώς παίρνω το λόγο και θα προσπαθήσω να κάνω φωναχτά ένα προβληματισμό, να σε εκφράσω αυτή την, τη σκέψη μου. Θέλω να ξεκινήσω ουσιαστικά μια συζήτηση στο πρόβλημα. Εγώ δεν κρύβω ότι έχω θετική στάση απέναντι στο φόρο. Υπάρχει και ένα θετικό, ε, όμως και ένα διοντολογικό θέμα και ένα τεχνικό θέμα και ένα πολιτικό θέμα γύρω από το φόρο. Η επιχειρηματολογία σας βασίζεται στο εξής. Εμείς στην Ευρώπη εφαρμόζουμε αυτό το φόρο μετά από μια σειρά από μελέτες. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι ο φόρος θα εφαρμοστεί και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και ότι θα γίνει παγκόσμιος φόρος τελικά αυτός. Τώρα, το ερώτημα που σας θέτω Ξέρετε πολύ καλά πόσο συνδεδεμένες είναι οι οικονομίες και πώς μπορούν οι διάφοροι ε, φορείς και παίκτες να επιλέξουν αγορές. Έχουν τεράστια δυνατότητα επιλογής. Ούτως ή άλλως υπάρχουν διαφορές μεταξύ της δικής μας ε, οικονομίας και των αναδυόμενων οικονομιών της Ασίας ή στην Αμερική όπου δεν υπάρχει αυτός ο φόρος. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξή. Και ούτω ή άλλω η βαθιά συζήτηση θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Αν αυτό ο φόρο δεν εφαρμοστεί, στις ασιατικές αγορές, στην αμερικανική αγορά, των Πολιτειών εννοώ, τότε μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ εναντίον μας. Και μπορεί να υπάρξει μεταγκατάσταση χρηματοπιστωτικής φύσεως οργανισμών, ιδρυμάτων κτλ. Γιατί όλη σας η λογική βασίζεται σε μία προϋπόθεση. Ότι αυτή είναι, λέτε, το πρώτο βήμα Προ τη γενίκευση σε παγκόσμιο επίπεδο του φόρου. Αυτή είναι η προϋπόθεσή σας, εκεί βασίζεται η επιχειρηματολογία σας και η πρόταση που μας κάνετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ δεν ε, θεωρώ ότι ανήκω στη δεξιά πτέρυγα. Εντάξει, το ξέρετε. Το ΕΛΚ είπε πάντα με μεγάλη πλειοψηφία ότι αυτός ο φόρος μπορεί να εισαχθεί μόνο εάν το κάνουν και άλλες χώρες παγκοσμίω. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να είμαστε και εκείνοι που θα προηγηθούν ίσως. Κάτι γίνεται εκεί στην ομάδα μας σχετικά. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις. Και θα ήθελα εδώ να στραφώ προς τον Επίτροπο. Θα πρέπει να ε, σας συμβουλεύσουμε βέβαια, αλλά εσείς πόσες πιθανότητες πιστεύετε ότι υπάρχουν το Συμβούλιο να εγκρίνει την εισαγωγή του φόρου αυτού γιατί χρειάζεται πλειοψηφία, ε, ομοφωνία έτσι δεν είναι. Και τέλος θα ήθελα να συγχαρώ για την τόλμη σας να υποβάλλετε αυτή την πρόταση. Γιατί όταν η Κομισιόν θέλει να περιμένει μέχρι να είναι σίγουρο ότι όλες οι χώρες θα συμφωνήσουν, δεν θα πετύχει τίποτα και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ καλό που υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα μετά από όλε αυτέ τις συζητήσει που είχαμε. Και μπορούμε έτσι να πούμε ξεκάθαρα να πούμε τι θέλουμε. Τέλος, είπατε ότι ε, αυτό τα χρήματα δεν θα συλλεχθούν από τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να είναι μια διεύρυνση των ιδίων πόρων. Αυτό είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Χουντή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Σεμέτα, αλλά επειδή από την ημερήσια διάταξη θα ήθελα να αξιοποιήσω την παρουσία του Επιτρόπου για τα θέματα καταπολέμησης της απάτης θα έλεγα για να μην βγάλω τη συζήτηση, ναι, κρατήστε με στο τέλος, δώστε στον κύριο Κλούτε την ερώτηση από την ομάδα μας και στο τέλος ας απαντηθεί γιατί είναι σοβαρή αλλά καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να διασπαστεί η συνέχεια των ερωτήσεων και ευχαριστώ πολύ. Αν μου δώσετε το χρόνο να πάμε και σε αυτό το θέμα για να διαξοπίσω την παρουσία του Επιτρόπου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος θα απαντήσει μετά και θα παρουσιάσει τα άλλα σημεία. Η κυρία Σουίνμπορν ε, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να περιορίσω αυτό που έχω να πω γιατί νομίζω πραγματικά ότι εδώ ε, έχουμε τεράστιες αυταπάτες. Δηλαδή, εάν νομίζετε ότι εμείς θα ξεκινήσουμε και μετά θα μας ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι, αυτό είναι πραγματικά κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί. Και εδώ πιστεύετε από την άλλη μεριά ότι τα κράτη-μέλη θα εισπράξουν χρήματα και θα τα δώσουν στην Ένωση περίεργο. 80% όλων των ε, συναλλαγών αυτή τη στιγμή γίνεται μεταξύ Λονδίνου και Φραγκφούρτη στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η συμβολή του ε, Ηνωμένου Βασιλείου στον ε, ευρωπαϊκό Προεπολογισμό θα εξαλειφθεί γιατί θα είναι τόσο σημαντική η συμβολή από το, το φόρο ή θα υπάρχει ο φόρος αυτός και θα εξαφανιστεί ο κόσμος ο χρηματοπιστωτικός από το Λονδίνο και θα πάει κάπου στην Ανατολή στις ασιατικές χώρες. Η αγορά της Ευρωβόντ είναι στο Λονδίνο από το 1963 λόγω των φόρων. Έχουμε επίσης αυτή τη σφυρική αγορά στο Λονδίνο λόγω του καθεστώτος το, του φορολογικού. Και πολλές συναλλαγές που γίνονται, γίνονται μέσω της αγοράς του Λονδίνου λόγω του αυτό είναι πιο βολικό και πιο οικονομικό. Εάν πιστεύετε ότι θα υπάρξει εδώ διεθνή συνεργασία, όχι. Αυτές οι συναλλαγές θα εξαφανιστούν. Δεν είναι ευρωπαϊκές συναλλαγές έτσι και αλλιώς, απλώς περνάνε από τις ευρωπαϊκές αγορές. Πραγματικά είναι τελείως ανόητο αυτό που ε, προτείνεται εδώ. Δεν λειτουργούν έτσι οι ε, χρηματοπιστωτικές αγορές πολύ λίγοι πληρώνουν αυτό το φόρο όπου υπάρχει στον εμβασίλειο που το ξέρω αυτό. Δεν θα λάβουν χώρα αυτά που ότι θα γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται οι πωλήσει αυτές εκτός το off με τις λεγόμενες spreading εταιρείες για να αποφευχθεί ακριβώς η καταβολή του φόρου. Λοιπόν, το να εισαγάγετε τώρα ένα κοινοτικό φόρο είναι τελείω ανόητο. Αν θέλετε να αλλάξει συμπεριφορά μέσω φορολογία, θα πρέπει ε, να δείτε ότι αυτός ο φόρος θα είναι πάρα πάρα πολύ μικρός. 209 δισεκατομμύρια ε, ευρώ το χρόνο ε, είναι οι συναλλαγές αυτές και πιστεύετε ότι θα εισπραχθούν φόροι πάνω σε αυτό. Όχι. Αν θέλει να εξαλειφθεί αυτή η αγορά από την Ευρώπη, το καλύτερο μπορεί να κάνετε να εισαγάγετε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκεγκούλτ. Well, first, uh, let me say uh, thank you to you. Πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσουμε. Για μένα, αυτή είναι μια ξεχωριστή μέρα, πραγματικά μια που δίνω τη μάχη με αυτό το φορά εδώ και μια εντεκαετία και όταν πήρα το πτυχίο μου και ξεκίνησα μια επιχείρηση τοπική με επιτυχία. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που επί 11 χρόνια τώρα προσπαθεί να ε, προωθήσει την υπόθεση αυτού του φόρου και για μένα να είναι εξαιρετική μέρα. ΑΤΑΚ λέγεται ο φορέας μας, μη κυβερνητική οργάνωση. Επομένω, είναι πάρα πολύ ξεχωριστή αυτή τη στιγμή και θέλω να σα ευχαριστήσω. Βεβαίω, είναι αυτονόητο ότι παγκόσμιο επιβάλλεται καλύτερα αυτό ένα τέτοιο φόρο. Κανεί δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, αλλά το μόνο θέμα είναι ότι αν δεν είναι δυνατόν να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, όπω και με άλλα μέτρα τα οποία θα θέλαμε να είχαμε επιβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο, μήπω καλύτερα να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Και αυτό το οποίο είπες ε, νομίζω ότι ήταν ε, αβάσιμο, λάθος, ε, δεν, δεν, δεν είναι ορθολογικό διότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που ακόμη εφαρμόζει φόρο χαρτοσύμου. Έχει κατόφλια και υπάρχουν ακόμα έσοδα περί το δισεκατομμύριο. Φόρο χαρτοσύμου έχει πάρα πολύ στενή φορολογική βάση. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό και θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να μπορεί να περιλάβει περισσότερο να είναι δικαιότερο. Όμω, οι άλλε χώρε δεν πρέπει να κάνουν το ίδιο. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί κατήργησε τον φόρο του η Γερμανία. Το έκανε για να ανταγωνιστεί καλύτερα το Λονδίνο. Γι' αυτό και λέγαμε την αθέμη του ανταγωνισμού στη δεκαετία του 90 και επομένω είναι σωστό τώρα εάν η Ευρώπη για να μπορέσει να έχει α, καλύτερο, πιο θεμητό σώρο ανταγωνισμού, ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Επίση σα διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν δυσμενεί επιπτώσει για την ανάπτυξη γιατί δεν ισχύουν αυτά τα οποία έλεγε η διαφάνεια ότι πάντοτε ο φόρος έχει αρνητικά σε επιπτώσεις τη της Αν κάτσετε και υπολογίσετε φόρο για μια ανάπτυξη αναχώρα, τότε θα δείτε ότι ο συσχετισμό είναι μηδέν. Γιατί εξαρτάται τι κάνει σε σχέση με το φόρο κάθε χώρα. Να, ένα υπέροχο παράδειγμα η Σουηδία, όπου έχουμε και υψηλό ρυθμό ανάπτυξη και υψηλό φόρου. Ε, είναι μια δημοκρατική επιλογή το κατά πόσο κανεί θέλει περισσότερου ή λιγότερου φόρου. Δεν είναι σχετικό με τον ρυθμό που τρέχει η ανάπτυξη. Τέλο, να είστε βέβαιος ότι εμείς θα σας στηρίξουμε και να είστε αυτό δεν θα γίνει διακύβευμα μεταξύ δεξιά και αριστερά. Επίση στη Γερμανία η Bundestag όλοι υποστήριξε αυτόν τον ε, φόρο και σε σχέση με το ότι θα επιβληθεί στην Ευρωζώνη στην αρχή. Επομένως, δεν είναι είναι θέμα κερδοσκοπίας ή όχι, και όχι δεξιά ή αριστεράς. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε ποιοι είναι οι τομεί που επιδέχονται φορολογία εύκολα στην Ευρώπη και ποιοι όχι στην Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνεται ορθολογικά συζήτηση. Χρειάζονται αυτά τα φορολογικά έξοδα. Η δε χρήση του. να μην πηγαίνει μόνο στον προπολογισμό των ευρωπαϊκό όπω γίνεται τώρα, αλλά θα πρέπει θα πρέπει να χρησιμοποιεί την κάτω πολεμάτα η, το έχει απαντού στον κόσμο και η κλιματική αλλαγή γι' αυτό και πάρα πολύ σωστό αυτό που κάνει αυτή ήταν η ρίζα της, ε, του αγώνα που δώσαμε δεν πρέπει να το ξεχνάμε Ευχαριστώ κύριε ε, Λούλη. Θα ήθελα καταρχήν να συμφωνήσω με εκείνους που σας συνεχάρισαν για το προσπάθεια αυτά. Πριν από ένα χρόνο τα ε, γερμανικά ΜΜΕ έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μάλλον επιφυλακτική όσον αφορά αυτού του τύπου το φόρο. Το είδα ξανά τώρα, το κοίταξα στην εφημερίδα και μου φαίνεται πάρα πολύ θετικό που ήρθατε σήμερα εδώ, μας παρουσιάσετε τη μελέτη αυτή και τοποθετηθήκατε ξεκάθαρα από αυτής. Από δική μου σκοπιά θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε και η κυρία Σφέρτσεν και ο κύριος Ρίγκολ η SPD, η Πράσινη και η Αριστερή στην ε, Γερμανική Βουλή, στον Bundestag, είναι ξεκάθαρα τοποθετημένοι υπέρ αυτού του φόρου, του λεγόμενου ΑΤΑΚ και πολλοί πολίτες επίσης το ζήτησαν με αιτήματα μέσω του διαδικτύου γιατί θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό. Και γι' αυτό αυτό που υποβάλλεται σήμερα είναι σύμφωνα με αυτό που πολλοί σκέφτονται τουλάχιστον στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ε, ερωτήσεις. Η Κέιτ Σφίντον αναφέρθηκε σε αυτό λίγο γιατί υπάρχει το θέμα της συνένεσης. Είναι κάτι που παρακολούσε και στο γερμανικά ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και ότι η Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον δεν είναι και πάρα πολύ ενθουσιώδη υπέρ τη πρόταση Από την άλλη μεριά μας απαιτεί το ομοφωνία. Ποια θα είναι η στρατηγική της Κομισιόν για να πετύχει εδώ την απαραίτητη ομοφωνία. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτά που είπατε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον φόρο αυτό για να δημιουργήσουμε μια νέα πηγή ίδιων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακριβώ και αυτό είναι από τα επίμαχα σημεία. Και στην Γερμανία, παραδείγματο χάρη, η γερμανική κυβέρνηση το εξετάζει πάρα πολύ επικριτικά. Δεν είναι δηλαδή κατά του φόρου, αλλά κατά του φόρου σαν έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια θα είναι η στρατηγική αντιμετώπιση. Τι θα κάνουμε ούτως ώστε να μην ξεκινήσει εδώ μια συζήτηση όπου θα συζητήσουμε θαυμάσια για ένα φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μέχρι που να χάσει κάποιο κάθε νόημα αυτή η συζήτηση. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος, αυτή η συζήτηση κάπως να αποτελματωθεί και το επιβεβαιώσα λίγο αυτό που διάβασα και στις εφημερίδες ε, στη Γερμανία προτείνεται, τα κράτη-μέλη ε, ότι μπορούν να προσθέσουν κάτι σε αυτόν τον φόρο και βέβαια ε, έχουμε πάλι το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών που τίθεται εάν τα κράτη-μέλη ζητάνε κάτι παραπάνω ανάλογα ή κάτι παρακάτω από το φόρο αυτό το κυρωτικό. Θα πρέπει λοιπόν να είναι απόλυτο το ύψος του φόρου αυτού, αλλιώς το αποτελέσμα θα ήταν αντιπαραγωγικό. Και τέλος, ε, για κάτι που είπε και της Πίντον, το ότι θα υπάρχουν μετατοπίσεις, αυτό είναι ένα επιχείρημα που ακούω για κάθε μέτρο και στην Γερμανία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ποτέ δεν έχω ξεκάθαρες αποδείξεις για κάτι τέτοιο. ότι υπάρχουν μετατοπίσεις επιχειρήσεων κλπ. είναι σαφές, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον σχετίζεται με αυτά τα θέματα. Και όταν συζητάω εγώ με επιχειρηματίες, ακούω ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι οι αγορές. Αντίστροφα, μπορούμε να πούμε, ας πούμε ότι αν θέλει κανένα μια περιοχή που να μην έχει κανένα φόρο, μπορεί να πάει στη Σαχάρα, που δεν έχει φαντάζομαι κανένα φόρο, αλλά δεν έχει καμία αγορά εκεί. Αυτό που ενδιαφέρονται οι επιχειρήσει είναι να πάνε σε μια αγορά. Όταν η αγορά αυτή είναι καλή, σωστή και αποδοτική, προτίθεται κάλλιστα να πληρώσουν φόρου οι επιχειρηματίε. Αυτό είναι γι' αυτό που άκουσα και ζητήσει και από πλευρά των επιχειρήσεων αυτών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να πάρω και εγώ το λόγο. Ο ως πρόεδρος, ως μέλος της Επιτροπής αυτής θα ήθελα και από τη μεριά μου να συγχαρώ τον Επίτροπο όχι για την ουσία της πρότατής του, αλλά για την αισιοδοξία του και την τόλμη του. Γιατί λέει ότι έχει μια νομική βάση, θα το δούμε αυτό. Αλλά είπατε επίσης ότι θα υπάρχει ενδεχόμενη φορολόγηση των μισθών και των πλημοδοτήσεων. Έχετε κάποια πρόταση για να φορολογήσετε τα εισοδήματα των πολιτών με ευρωπαϊκό φόρο. Μια ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Θεωρείτε ότι μπορείτε να φτάσετε σε εισοδήματα της τάξης των 200 δις. Αυτό από κάπου θα πρέπει να προέρθουν βέβαια τα κράτη-μέλη φορολογούν τις τράπεζες τώρα. Εάν λοιπόν θα πρέπει να πληρώσουν αυτό το συμπληρωματικό φόρο, θα έχουν μικρότερο εισόδημα οι τράπεζε αυτές για να φορολογηθεί από τις χώρες τους. Δεν μπορεί κανένας να του φορολογήσει διπλά έχετε μελετήσει τις επιπτώσεις αυτές, τις ενδεχόμενες απώλειες των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά το εισόδημα που έχουν αυτή τη στιγμή από την φορολογία ε, επί του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτά. Θα πρέπει να είμαστε νομίζω πολύ προσεκτικοί. Αυτές οι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγές που δεν θα λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Πράγμα πολύ εύκολο. Δεν θα αποδίδουν εισόδημα. Προφανώ. Αναφερθήκατε στον κίνδυνο που υπάρχει σχετικά με την πτυτικότητα κλπ. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Πρόσφατα ε, υποδεχτήκαμε τον κύριο Τρισέ εδώ πριν από δύο εβδομάδες και εγώ του υπέβαλα πάλι μια ερώτηση γιατί η Κομισιόν μόλις είχε πει ότι είναι υπέρ αυτού του φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ως ιδίους πόρους. Και εάν υπάρξει, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ίδιος πόρος αλλά ο κύριος Τρισέ είπε ξεκάθαρα ότι θεωρεί ότι πρόκειται για σφάλμα. Εάν αυτός ο φόρος ε, δημιουργηθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ συζήτησα με κάποιον από τους από τους μεγάλους ε, ε, τραπεζίτες της Ευρώπης και μου είπε μπορεί να είσαι υπέρ. Δεν θα πετύχει ποτέ. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το, όνομά σας. Αν είσαστε πρόεδρος μπορείτε να έρθετε να με αντικαταστήσετε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε το λόγο. Έχετε το... Κύριε Επίτροπε, όπως και οι συνάδελφοί μου, χαιρετίζω τα αποτελέσματα τα προκαταρτικά αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου. Έχω δύο τεχνικές ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ότι η επίπτωση είναι το πιο δύσκολο πράγμα να αξιολογηθεί. Ε, το θέμα της μετατόπισης του φόρου. Και ανάλογα με την ελαστικότητα, δεν είναι αυτός που μοιάζει να πληρώνει αυτός που θα φέρει το τελικό φορολογικό βάρος. Διερωτώ αν τα αποτελέσματά σας δείχνουν αν τελικά τα υψηλά εισοδήματα θα φέρουν αυτό το βάρος ή μήπως τα χαμηλά εισοδήματα, οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Επίσης, τα χρηματοπιστωτικά κέντρα που κάνουν αυτές τις συναλλαγές, αυτά θα φέρουν το βάρος ή οι κάτοχοι των ομολόγων και των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων και προϊόντων. Δεύτερο ερώτημα. Για τον φόρο που είναι φόρο συναλλαγών. Θα θυμάστε το φόρο πωλήσεων και τον φόρο τον ΦΠΑ δηλαδή. Που είναι, ο φόρος πωλήσεων είναι ένας φόρος συναλλαγών. Φορολογεί λοιπόν κάθε συναλλαγή αυτός ο φόρος πωλήσεων με έναν τρόπο που βοηθάει τα χρηματοπιστωτικά όργανα ή τις εταιρείε που κάνουν τις συναλλαγές μέσα στην εταιρεία, γιατί δεν εκτίθεται στο χώρο αλλά τις μικρές εταιρείε που ουσιαστικά τελικά δεν κάνουν αυτές τις συναλλαγές άμεσα, αλλά ε, εκχωρούν τις αρμοδιότητες, τελικά φέρουν το βάρος. Αυτό ισχύει, το, αυτό το πράγμα που ισχύει για το φόρο των πωλήσεων ισχύει και για το φόρο αυτό των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα δώσω πολύ σύντομα το λόγο στον κύριο Φαγιό, σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο Τελειώνουμε με την ερώτησή σας και θα απαντήσει ο Επίτροπος για το φόρο αυτό των χρηματοπιστωτικών σταλών και έχουμε και άλλο σημείο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός. Έχω μια τεχνική ερώτηση. Θέλω να καταλάβω τη μορφή για την ίσπραξη αυτού του φόρου. Τι θα συμβεί ακριβώς οι φορολογικέ τοπικές υπηρεσίες θα εισπράττουν ή θα δημιουργήσουμε μια νέα ε, υπηρεσία που θα εισπράττει. Θα λάβουμε επίση υπόψη μας το κόστος που συνεπάγεται η εισπράξη αυτού του φόρου. Υπάρχει πάντα ένα κόστος κάτι την εισπράξη. Θα το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κάποιες ήταν τεχνικές ερωτήσεις, αμυγός τεχνικές. Όπως σας είπα, ακόμη επεξεργάζομαστε την πρόταση. Και τα τεχνικά ερωτήματα χρήσιμο θα ήταν να τα συζητήσουμε σε μια μεθεπόμενη συζήτηση, σε τεχνικό επίπεδο όμως. Και όλα αυτά τα τεχνικά ερωτήματα θα μπορούσαμε εκεί να τα απαντήσουμε. Γιατί τώρα αν μπω σε πολλές λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως, θα μας πάρει μάλλον πολύ χρόνο. Προτείνω λοιπόν να οργανώσουμε Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρόταση, μια τεχνική συζήτηση, μια τεχνική ενημέρωση με τις υπηρεσίες της Κομισιόν και να μπούμε στα συγκεκριμένα τεχνικά ερωτήματα της πρότασης. Uh, uh, uh, global, Τώρα για τα πιο παγκόσμια θέματα, για τα χρηματοπιστωτικά κέντρα, για αυτό που είπε η Αγγλίδα συνάλληφος για το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, πώς μπορεί να επηρεάσει τις άλλες χώρες. Είναι ενδιαφέρον να σας πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεταξύ αυτών των χωρών που έχει τέτοιο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όχι μόνο αυτό το τέλος χαρτοσύμου για τις ε, μοτοχές ή τους τίτλους, αλλά έχει και φόρο στα παράγωγα, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στα παράγωγα. Και παρόλα αυτά, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένα μείζον χρηματοπιστωτικό κέντρο στον κόσμο. Τώρα, για την Ασία, η Ταϊβάν, ας πούμε, έχει τέτοιο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και είναι επίσης ένα από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα στην Ασία. Η Ελβετία, επίσης, έχει ένα τέτοιο φόρο συναλλαγών και για τους τίτλους και για τα ομόλογα διαφορετικό φόρο ανάλογα με το μέσο, αλλά είναι ένας εγχώριος φόρος, τοπικός φόρος, που είναι, έχει χ ε, φορολογικό συντελεστή και, έχει, και έχουμε άλλο φορολογικό συντελεστή ψ για τις α, ε, ξένες συναλλαγές. Έχουμε και άλλα παραδείγματα τέτοιων φόρων. Και παρόλα αυτά, οι χώρες αυτές που επιβάλλουν αυτούς τους φόρους παραμένουν μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Και τα έσοδα από αυτούς τους ε, φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι και τόσο ε, χαμηλά όσο είπατε. Μιλάμε για δις ευρώ, έτσι, ή δις τερλίνες. Μιλάμε για μεγάλα ποσά. Για μεγάλα έσοδα από τους φόρους αυτούς. Τώρα για τα χρηματοπιστωτικά λοιπόν κέντρα και για το ποιος θα πληρώσει το φόρο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν η συναλλαγή γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Γερμανία ή στη Γαλλία, που είναι τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτές οι συναλλαγές εκτελούνται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αυτών των χωρών. Γι' αυτό λοιπόν αναλύουμε τη δυνατότητα να βάλουμε την αρχή της φορολογικής κατοικίας ή έδρας που θα μας επιτρέπει να εισπράττουμε το φόρο στη χώρα όπου το ίδρυμα αυτό δραστηριοποιείται. Αν παραδείγματος έχουμε ένα αυτιακό ίδρυμα ας πούμε, που κάνει μια συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συναλλαγή αυτή μπορεί να φορολογηθεί στην Αυστρία και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εισπράξει η Αυστρία, λέει, οι αυστριακές αρχές και όχι οι αρχέ του Βασιλείου. Αυτό ε, τώρα είναι λεπτομέρειε τη πρόταση. Συμφωνώ πλήρω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί και εδώ απαντώ στην κυρία Λούλινγκ. Είμαι συνετός εγώ ίδιο. και θα συνεχίσω προ αυτή την κατεύθυνση με μια τέτοια πρόταση. Τώρα για τον κύριο Τρισέ, στις παρατηρήσεις του, α, μ' άρεσε η δεύτερη παράγραφος, όπου είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να είμαστε συνετοί όταν εισάγουμε ή κάνουμε βήματα για την εισαγωγή ενό φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε νοσιακό επίπεδο. Δεν είπε ότι είναι αδύνατο. Είπε ότι πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά απλώ. Εκτός μικροφώνου ο διάλογος. Συμφωνώ με την άποψη του πάντως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να σχεδιάσουμε πολύ προσεκτικά το φόρο. Γι' αυτό ακριβώς σκεφτόμαστε τα επίπεδα του φόρου. Και οι στελεστές είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Λαμβάνουμε υπόψη μας δηλαδή ότι είναι μια ευρωπαϊκή λύση αυτή και όχι παγκόσμια λύση. Αν όμως υπάρξει παγκόσμια συμφωνία, φυσικά αυτοί οι στελεστές μπορεί να αυξηθούν γιατί τότε ο κίνδυνος μετατόπισης ή με την κατάσταση, ας πούμε των Ιδρυμάτων δεν θα είναι σημαντικός. Όλα αυτά τα στοιχεία τα επεξεργαζόμαστε. Το θέμα της αντίδρασης του Συμβουλίου τώρα. Και για πώς θα αντιδράσει στην πρόταση εισαγωγή αυτού του φόρου και υπαγωγής του στους ίδιους πόρους. Πιστεύω ότι μπορούμε να προτείνουμε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα φορολογικών συντελεστών ω συνεισφορά στους ίδιου πόρους και να αφήσουμε την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ανέβουν να ανεβάσουν το συντελεστή και η διαφορά να πάει στο, στον εθνικό κορβανά. Τότε η συνεισφορά του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος θα μειωθεί για τα κράτη-μέλη. Και αν βάλουν και κάτι παραπάνω, θα μπορούσαν να εισπράξουν περαιτέρω έσοδα για τους προπολογισμού τους, λοιπόν. Και επομένως θα έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά για φορολογικούς σκοπούς, ε, ειδικά όταν φορολογούμε το χρηματοπιστωτικό τομέα. Τώρα έχουμε διάφορα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν αναπτύξει τη δική τους προσέγγιση για τη φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και ακόμα και μικρές διαφορές σε αυτή την προσέγγιση δημιουργούν προβλήματα διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης, διάφορες δυσκολίες, εν με την εφαρμογή των φόρων αυτών. Τώρα για την νομική βάση. Όταν μίλησα για την νομική βάση, λέω, εννοούσα ότι με βάση την ανάλυση μας προκύπτει ότι και ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή και ο φόρος χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων μπορεί να βασιστεί στο άρθρο 113 της συνθήκης. Μπορεί να βασιστούν και οι δύο. Δεν θα φορολογήσουμε επίσης άμεσα τους πολίτες. Ο φόρος δραστηριοτήτων θα αφορά τα έσοδα και τις απολαβές των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα φορολογεί τις συναλλαγές και ούτως ή άλλως θα, υπάρξει μια, θα υπάρξουν αντισταθμίσεις στο φορολογικό ε, τομέα. Κάτι άλλο ενδιαφέρον Με βάση τις εκτιμήσεις μας, το 85% όλων των συναλλαγών εκτελούνται μεταξύ φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα, παραγόντων και φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε όταν μιλάμε για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Έχει τεράστιο μερίδιο στο, στις συνολικές συναλλαγές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Και το μερίδιο των συναλλαγών ε, εκτός των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων, δηλαδή των πολιτών Φερρυπίν κτλ, είναι πολύ περιορισμένη η συμμετοχή. Θέλουμε λοιπόν να σχεδιάσουμε το φόρο με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να τον περιορίσουμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι στους πολίτες και λοιπούς. Τώρα, η πρώτη πρέπει να περάσει πάμε με ομοφωνία. Υπήρχαν πολλέ ερωτήσει σχετικά με το θέμα αυτό. Πώ θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή τη στάση του Συμβουλίου. Έχω ήδη απαντήσει για το θέμα του Συμβουλίου, αλλά μην ξεχνάμε και είναι σημαντικό οι ευρωβουλευτέ να πάρουν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε και να την χρησιμοποιήσουν στα κράτη-μέλη, να την προωθήσουν να προωθήσουν τις ιδέες αυτές και την προσέγγιση. Ο ρόλος επίσης των πολιτών είναι πολύ σημαντικός. Και με βάση τις τελευταίες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου φαίνεται ότι το 61% των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζουν την εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου σε ενωσιακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα θετικό πλαίσιο, ένα θετικό περιβάλλον γύρω από αυτήν την ιδέα. Τώρα για το Συμβούλιο. Όταν οι αρχηγοί της Ευρωζώνης συζητούσαν το πακέτο, υπήρχαν και τα σημεία όπου τα μέλη της Ευρωζώνης κάλεσαν την ε, Κομισιόν να εισαγάγει και να διερευνήσει το επίπεδο τη εισαγωγή αυτού του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη σε αντιδιαστολή με την Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να το ψάξουμε εμεί. Μα κάλεσε το Συμβούλιο να το κάνουμε. Πιο συγκεκριμένα, μάλλον τα μέλη τη Ευρωζώνη. Όπω με κάθε πρόταση όμως για φορολογία, χρειαζόμαστε ομοφωνία. Θα πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά από όλους μας, από την Κομισιόν, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ μαζί με τους συναδέλφους μου, αλλά και από αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Βέβαια, έχω υπόψη μου βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Υπάρχει άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ε, η καταπολέμηση της απάτης ο κύριος Χουντής εδώ. Μπορείτε να θέσετε γρήγορα το ερώτημά σας κύριε Χουντή για την καταπολέμηση απάτης. Γιατί ε, στις 4.30 πρέπει να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πάλι. Η ερώτηση έχει σχέση με την αρμοδιότητα του Επιτρόπου που έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας αρμοδίου για τα θέματα καταπολέμησης της απάτης και ήθελα να του κάνω ορισμένα πολύ απλά ερωτήματα. Υπάρχουν μια σειρά σκάνδαλα, οικονομικά σκάνδαλα και σκάνδαλα διαφθοράς που αφορούν μεγάλες εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πλειοψηφία γερμανικές. Αναφέρομαι στη Siemens, στη Ford Motors, στη MAN και ούτω καθεξής. Και έχουν σχέση με καταγγελίες ότι προκειμένου να πάρουν έργα και δημόσιες προμήθειες δωροδοκούν εθνικούς αξιωματούχους. Δυστυχώς κύριε Επίτροπε αυτά έχουν έρθει στην επιφάνεια από δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ η αίσθηση και από στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου είναι ότι η Επιτροπή διακρίνεται από μεροληψία ή και ασυλία. Ερωτήσεις που έχω κάνει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι σχετικά με το τι κάνετε διότι πρόκειται περί των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογούμενων, οι απαντήσεις δεν είναι σαφείς. Σας ερωτώ λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Θα σας απασχολήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι και η Κομισιόν, εσείς αλλά και ο προκάτοχός σας έχετε ευθύνη για αυτό το θέμα. Αληθεύουν αυτό που λέγεται ότι υπάρχει μεροληψία επειδή είναι γερμανικές εταιρείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσει ο κύριος Επίτροπος. Βέβαια. Η απάτη είναι θέμα του χαρτοφυλακίου. Και βέβαια ε, ε, για την απάτη έχουμε τη φορολογική απάτη, για την άλλη μεριά έχουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση και τις σχετικές απάντες. Πάρα πολύ σκληρά προσπαθούμε να καλύψουμε και την μεν και την δε απάτη και αναπτύξαμε μια στρατηγική κατά της απάτης. Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε σημαντικά το προστάσιο κατά της απάτης και δουλεύουμε και προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Εντείνουμε τις προσπάθειες. Ε, γίνονται επίσης επιχειρήσεις επιτόπου, συγκεκριμένες, στοχοθετημένες για διαφορετικά είδη απάντηση και ενδεχομένω στον τύπο. Έχετε διαβάσει για μια σειρά περιπτώσεων που δημοσίευσαν, δημοσιοποίησαν τα μέσα μας ενημέρωση. ενημέρωσης μια που τα θεσμικά όργανα ε, προχωρούν σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε είναι και θέμα όλα και τη εντολή τη. και επομένω έχει αναλυθεί δράση Εκτό από τη στρατηγική κατά τη απάτης επίση. Έχουμε ένα πρόγραμμα δραση για τα ανατολικά σύνορα για λαθρεμπόριο. Τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά. Δεν πρόκειται για εγκλήματα που αποστερούν σημαντικών εισοδημάτων την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ζητηθεί αυτό στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Κόντου και σας καλώ να συμμετάσχετε. Τώρα έχουμε μια νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ. Τα θέματα απάτης είναι κορυφαία προτεραιότητα. Και ακριβώς προτίθεμε μέχρι τέλους του έτους να έχουμε προχωρήσει. Ως πρώτο τώρα τις ε, επιχειρήσεις. Ξεκινήσαμε το Eurofisk. Με στόχο να ε, διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών τα κράτη-μέλη θα καταπονημήσουν πιο αποτελεσματικά την ε, απάτη με τον ΦΠΑ. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως υπάρχουν και προτάσεις για αυτή τη νέα στρατηγική που περιλαμβάνει και στοιχεία καταπονήμησης απάτης. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μακρά βέβαια συζήτηση όσον αφορά τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Γιατί δεν μπήκαμε σε θέματα άλλης φορολογίας. Και αν θέλετε για τα υπόλοιπα θέματα που θα μπορούσατε να μας μιλήσετε, μπορείτε να μας ε, γνωστοποιήσετε απόψε σας εγγράφους. Και για να μπορούν να έχουν και κάτι να διαβάζουν στην παραλία οι συνάδελφοι. και να είμαστε έτοιμοι για μετά. Σα ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για τα όσα μα είπατε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Άρα, περιμένουμε την νομοθετική πρόταση τώρα. Το φθινόπωρο. Πάντω, ευχόμαστε. Καλές διακοπέ, και ευχαριστούμε που ήρθατε. Επίτροπο. Να ευχαριστήσω αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ τους ξέρουμε βουλευτές και βεβαίως θα σας απαντήσουμε γράφω όσον αφορά την πρόοδο αυτών των σημαντικών θεμάτων. Και εσείς ε, στη συγκύρια και τα Τάισεν επίσης ξέρω ότι περιμένετε πώς και πώς να συγχυστεί για αυτά τα θέματα η συνεργασία μας. Και εγώ θεωρώ ότι είναι φύση σύμμαχό μα το Κοινοβούλιο. Μαζί θα προωθήσουμε αυτά τα θέματα. επομένω, σα ευχαριστώ. Σα εμεί σα ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα λάβει το λόγο ο Αντιπρόεδρος, γιατί πρέπει εγώ να προβώσω σε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με το διορθωτικό στην έκθεση Σμιτ. Όλοι Σμιτ. Κατόπιν της που έγινε στις 5 Ιουλίου σαν αφορά την έκθεση Σμιτ για την ε, την οδηγία εκείνη έχουμε ένα έγγραφο διορθωτικό έγγραφο όσον αφορά ε, αυτό το σχέδιο κειμένου σήμερα με το άρθρο 261 του κανονισμού μας έχετε όλοι λάβει την Παρασκευή αυτό το έγγραφο, το Ιουλίο. Εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, τότε αυτό το διοικητικό έγγραφο θα υποβληθεί στο σώμα. Στην πρώτη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Και αν δεν υπάρχει ένσταση από πολιτική ομάδα ή από 40 βουλευτές, τότε θα θεωρηθεί ότι υπερψηφίζεται αυτό το διορθωτικό ιδάλλως θα τεθεί σε ψηφοφορία. Θα ενημερωθούν τα μέλη στο πλαίσιο του τριμμένου διαλόγου αύριο από την πρόεδρο. Κάτι άλλο το που θα πρέπει να το εγκρίνουμε. Πρόκειται για το σχέδιο χρονοδιαγραμμάτων των συναντήσεων μας για την επόμενη χρονιά. Κύριε Ραμπέρ, έχει λόγο. Θέλω κάτι να ζητήσω, κάτι να πω όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας αλλά και του ιδιωτικού επίπεδου. Είπαμε ότι αρχές Ιανουαρίου δεν θέλουμε να έχουν ψηφορήσει στην Επιτροπή μας. Αυτό το λέω στην ε, γραμματεία, να μην προβλέπονται στην αρχή της χρονιάς για να μπορούμε να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας με διακοπές. Πρόεδρος, ναι επιβεβαιώθηκε 9 Ιανουαρίου δεν θα γίνουν ψηφοφορίες. Τώρα θα ψηφίσουμε. Τεχνικέ απαιτήσει για τις μεταφορές πίστοση. Άμεσε χρεώσει. Σε ευρώ. Τροποποίηση του κανονισμού 924 2009 η κυρία ήταν η κυρία Εσαγιά. Δεν είναι εδώ. Α, Α εδώ είναι. Έχετε εδώ την κατάλληλη ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Συγγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα ε, τον ε, συμβασμό Λαϊκού Κόμματος Έλλη και Πρασίνων υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο 16. Φορά το 1-1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το 124. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 εισηγείται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συνδεσμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 εισηγείται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 137 έχει αποσυρθεί, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 της ίδρυας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτα άσου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε, θήτα γιώτα ζ γιώτα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 L λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M λατινικό είναι χωριστή ψηφορία το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχο ψηφορίας. Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Λαμπέρ. Εκτός μικροφώνου και ο Τι ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρο. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρα. Το δεύτερο τμήμα. Πέρα. Αποτέλεσμα. 28 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ράμπερ, κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορείτε να μας τα πείτε στα Λουξεμβουργία. Τα Λουξεμβουργιά να πούνται ακόμη τόσο συχνά. Ε, λυπάμαι δεν είναι γλώσσα, επίσημη γλώσσα εργασία. Θα ήθελα πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τα λέει στα να το ίδιο. Λυπάμαι δεν μπορώ. Και ο μιλάει Ισραήλ. Ναι, υπέρ, κατά, όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά να νομίζω να ελέγξουμε καλύτερα την 163 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι Πέρασε. 29 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές. Α, όχι, έχει καταπέσει. 16. Α, συγγνώμη, ναι, ναι, έχει καταπέσει πράγματι. Δεν πειράζει. 164. Δεν είναι τραγικό, λέει ο ήταν τη ΙΜΚΟ. 164 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 168. Να ελέγξουμε. Ευχαριστώ. Για την 164 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 164 του κ. Φέρμπερ. Ψήφισατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 100 κατά. Πραγματικά απερίφθη. Καλά είπα. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 169. Vous avez tous voté. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 38 υπέρ 7 κατά. Συμβαστική π. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξω. Άρχιψη ψηφοφορία. Πέρας. 6 υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177 επεσύρθη. Συμβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Ελέγξουμε. Συμβαστική του Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ 20 κατά. Απαραίτητα. 183 υπέρ κατά. Αποχές. Απαραίτητα. 185 υπέρ κατά. Αποχές. Απαραίτητα. 52 υπέρ με συγχωρείτε, διακόπτεται από την γραμματεία. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστά. Αφού η συμβαστική απερίφθη, πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία τις άλλες τροπολογίες από την οποία αποτελεί το. 178 γκοζές υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κύριε Γκοζέ, είσαι υπέρ της τραπολογίας ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, να εξε... ακολουθήσουμε τον κατάλογο της ψηφοφορία σιγά σιγά και να εξηγείτε κάθε φορά στους συναδέλφους τι ψηφίζουν. Μάλιστα. Είχαμε ψηφίσει πάνω στην τροπολογία ΚΟΥ, συμβαστική, η οποία απερίφθη. Νομίζω ότι ίσως παραβιάστηκα. Δεν ξέρω. Θα ξαναψηφίσουμε πάνω στην βαστική τροπολογία. Όχι, όχι, απερίφθη η συμβαστική. Αλλά μετά μπερδευτήκαμε. Ναι, ναι. Θα ξαναρχίσουμε με τη ζευγορία για τη συμβαστική. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Μπούλαμ. Ήταν σαφές. Μα αφού ήταν σαφές qui est pour Μα ακούστε, υπήρχαν συνάδελφοι που δεν είχαν κατά. Μα ψηφίσαμε ηλεκτρονικά. Θα ξαναψηφίσουμε τη συμβαστική κου γιατί δεν ήταν σαφές. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Μα ψηφίσαμε ηλεκτρονικά πρόεδρε. Δεν μπορεί να υπάρχει λάθος απερίφθη συμβαστική ηλεκτρονικά. Κρίμα. Νομίζω ότι εγώ ίσως παραβιάστηκα. Δεν ξέρω. Και όλοι μέσα στην δεν είχαν καταλάβει τι ψηφίζαμε. Ναι, προχωρείτε γλίγορα και δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε. Μα γι' αυτό θέλω να επαναλάβω την ψηφοφορία, ακριβώς. Τώρα χάνουμε χρόνο. Δεν θέλετε να ψηφίσετε πάνω στο κου γιατί απερίφθη. Κρίμα όμως, πολύ κρίμα. Γιατί κατέρευε σημαντική προσπάθεια ΣΥΤΕΣ. Μα πρόεδρε, γιατί φοβού, φοβάστε δηλαδή μια επαλήθευση. Δέκα λεπτά συζητάμε εδώ κάτι δεν πάει καλά νομίζω. Γιατί όλοι αν με τον ίδιο τρόπο, τελείωσε. Λοιπόν, λέει η θα επανεξετάσουμε τη συμβαστική Q. Άκρη ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μα τι ψηφίζουμε ρωτάει κάποιος. Για την συμβαστική Q ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ωραία. 16 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Άρα πραγματικά απερίφθη. Αλλά επειδή απερίφθη συμβαστική, κοιτάξτε, αν κάποιοι δεν είχαν καταλάβει περί τίνο πρόκειται, εντάξει ψηφίσαμε ξανά το ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία. Απερίφηση συμβαστική. Και ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 178. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές Υπέρ της 179 κατά απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Μπούλμαν. Πρόεδρε, θα να συζητήσω στην ομάδα μου σύμφωνα με τους νέους όρους να υπερψηφίσουν τώρα την 182 εναντίον με αυτό που πάει στο κατάλογο της ψηφοφορίας. Δεν ξέρω το κατάλληλο η ομάδα σας κύριε Μπούλβαν. Λοιπόν, 182 υπέρ κατά Υπέρ της 182 παρακαλώ. Κατά. Για να ελέγξω. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 182. Άρχεται. Πέρασε. 18 υπέρ 18 κατά. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι πολύ σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ 18 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική R. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τοπολογία 196. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά απορρίπτεται νομίζω θέλετε να ελέγξουμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 53 ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ 19 κατά Απερίφθη. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 20. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίες. 20 υπέρ 15 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 210. 210 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Άρχη ψηφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. 18 υπέρ 19 κατά. Απορρίπτεται. 211 υπέρ κατά έλεγχος. Ψήφισαν όλοι πέρες ψηφοφορίες. 18 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. 21. Ήμκο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 21 ΙΜΚΟ. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 25 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. 22. ΙΜΚΟ Υπέρ. Ψήφισαν όλοι. όχι υπέρ της 20.2 20.2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστικές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 αποσύρθη Α, ναι, επεσύρθη. 56 λοιπόν, υπέρ. Κατά. 56, έξι, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 217, απεσύρθη. 57 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός 218 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 21 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 καταπίπτει 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ α κατέπεσε 66. 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Α, κατέπεσε, κατέπεσε, κατέπεσε. 25 υπέρ. Α, κατέπεσε και αυτή. Ωραία. Ο κατάλογο που έχω στα χέρια μου δεν είναι πολύ σαφή. Συμβαστική U, υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Κοσμίωση V, υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 27, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 27. Έλεγχο ηλεκτρονικό για την 27. Ψήφισαν όλοι. πέρα. 19 υπέρ 18 κατά. Εγκρίθηκε. 228 υπέρ. Κατά. χες εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α, εγκρίνεται. Συμβαστική X. Χ. Α, όχι ένα λεπτό. Il n'y a pas de... C'est tombe, Alexa, le, mais euh, nous sommes déjà plus loin. Ah, ah, ah η 72 δεν είχε καταπέσει. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβαστική W την ψηφίσαμε. Συμβαστική ε, 74 υπέρ. Όχι, όχι, τη συμβαστική χ ξεχάσαμε. Συμβαστική χ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία του εισηγητή που είναι γραπτή εδώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ή 75 κατέπεσε, 76 λοιπόν υπέρ και 29 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 ταυτόσημοι 78 και 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 και 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 και 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική υψηλών γκρέκ υψηλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά Διακόπτη πρώτα. Στην 84 έχουμε φτάσει. Μετά τη συμβαστική Y ε, περνάμε στην 84. Α, ο μπλοκ θέλετε. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Λοιπόν, 84 Μέχρι πού? Μέχρι 93. Ναι, αλλά στο 94. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 237, υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ζήτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ζήτα α συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ZC στα γάμα σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα χωρίς την όρο υποχρεωτικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, αυτή τη λέξη mandatory υποχρεωτικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ZD, ZD, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 108, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 108. 108 ε, λέει πρόεδρο του κυρίου Χουντή. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 21 υπέρ 17 κατά. Εγκρίνεται. Το 2 υπέρ κατά. Για να ελέγξουμε. 2 ημκο. Le vote est clos. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 25 υπέρ, 12 κατά. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. 109, 110 και 3. Είναι ταυτόσημα. Και η 11 λέει η πρόεδρος. Α, όχι 11. 109, 110 και 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Να ελέγξουμε. ηλεκτρονικό έλεγχο για τι τρει αυτέ τροπολογίε. Πέρα. 21 υπέρ 16 κατά. Εγκρίνονται. Έντεκα του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε Le vote est για την 112. 20 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική ζητά ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 115. Έλεγχος για το ΖΕ. Παρακαλώ. 16 υπέρ ή 20 κατά. Άρα απερίφθη. Άρα θα ψηφίσουμε τα 113 υπέρ. Ναι, αφού κατεψηφίσει η συμβαστική θα πρέπει να ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Άρχισε φορέ. Tout Ψήφισαν όλοι. 14 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ZF. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ζέτσι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 απεσύρθη ή 15 υπέρ. Α, ξέχασα μία συμβαστική. Ζετάς. Ζητάει τα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Α, στο κείμενο πρώτα. Ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι υπέρ της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 3 κατά. 10 αποχές. Το νομοθετικό ψήφισμα. Τώρα πάλι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 2 κατά και 13 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάγια, θέλετε το λόγο? Έχετε το λόγο. Yes, uh, my... Κυρία Πρόεδρε, δέχτηκε την έκθεσή μου η Επιτροπή. Ζητώ λοιπόν την άδειά σας να ξεκινήσω τον τριμερή διάλογο πάρα αυτά, ούτως ώστε να περάσει σε πρώτη ανάγνωση, αν γίνεται. Ζητώ λοιπόν την άδεια της Επιτροπής για να προχωρήσω στον τριμερή διάλογο, στον τρίλογο δηλαδή. Ε, Ακούσατε τι είπε η συγκήτρια. Συμφωνείτε με την πρότασή σας να ξεκινήσει πάρα αυτό ο τρίλογος. Θέλετε να ψηφίσουμε. Ο κύριο Γκώστας δεν συμφωνεί. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε επί της πρότασης της εισηγήτρια να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Tout Ψήφισαν όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 10 κατά. Μπορείτε να ξεκινήσετε λοιπόν τον τριμερή διάλογο, κυρία μου. Και σας ευχόμαστε κουράγιο και επιτυχία βέβαια. Euh, Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Πάμε τώρα στο σημείο 6 διαδικασίες αφαιρεγγιότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις ε, επιχειρήσεις. Αν μου δώσετε λοιπόν τον κατάλογο ψηφοφορία, θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε το συμβασμό α, α ποιος είναι υπέρ, με μια τροποποίηση, ε, την, τεχνική τροποποίηση που είδατε όλοι σας. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, υιοθετείτε. Συμβασμός Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός Σ. Γ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός Δ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Πάραχο 3. Χωριστές ψηφοφορίε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. παράχως 5. Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. Πάραφος 6, ε, τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Συμβασμός ε, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Συμβασμός ε, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Παράγραφος 7, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Και τώρα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 0 ε, ψήφι κατά, 0 αποχές, συγχαρητήρια. Συγχαίρουμε την απούσα πρόεδρό μας. Θα της πούμε όμως τα καλά νέα. Και τώρα πάμε στο σημείο 7, τροποποίηση των οδηγιών 89 κάθετος 666 και των υπολείπων για την διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρών καθώς και των μητρών εταιριών. Ε, ο συντάκτης είναι ο κύριος Μάρτιν. Ξεκινάμε το πρώτο άρθρο, τροπολογία 45. Α, όχι, αποσύρθηκε διορθώνει πρόεδρος. Τροπολογία 46, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετειτε συμβιβασμο Συμβιβασμός 1α. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Υιοθετείτε. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε on block. 15, 16, 17, 18. Υπέρ. Κατά. Υπέρ, υπέρ, υπέρ. Κατά τώρα, αποχές, υιοθετείτε. 48, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 49, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Υπάρχει μια νέα. Ψηφίζουμε τις κατεξιότητες πράξη 19, 20, 21, 22. On block. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Και τώρα το ίδιο πάλι. On block, 24, 27, 28, 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Και τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την 25 του εισηγητή. Όχι. Έτσι μου είπαν εδώ. Επιμένουν. Διαφωνούμε. Να ψηφίσουμε, λοιπόν. Γιατί το... η ομαδική ψηφορία δεν καλύπτει 25. 25 υπέρ, κατά... Την 25, έτσι. Πρέπει να ψηφίσουμε την 25. Θα μας συμφωνήστε να τα βρει, βρείτε τα. Ψηφίζουμε την 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβιβασμός ΑΒ υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι υιοθετείται, αλλά στο επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Για το Α. ΑΒ, έτσι. Ψήφισαν όλοι. τη ψηφοφορία 24 υπέρ 14 κατά. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 33 υπέρ. Κατά. απόχέ, Υιοθετείτε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό α. Γ. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Υιοθετείτε. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το επαληθεύσουμε. Το 39. Πέρας προφορίας. 8 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό α. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Υιοθετείτε. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 8. Υπέρ. Ελέγχουμε. Το 43. Το ελέγχουμε το 43. Πέρας 15 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, εποχές, υιοθετείτε. 9 υπέρ, κατά, εποχές, υιοθετείτε. 10 υπέρ, κατά, εποχές, υιοθετείται. Συμβασμός Β. Το 10 θέλετε να το επαληθεύσουμε. Ναι. Ψηφίζουμε το 10. Πέρας προφορίας. Τώρα. 25 υπέρ, 13 κατά. Υιοθετείτε. Συμβασμός Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Το κείμενο. Υπέρ. Ηλεκτρονικά το ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ας τους λίγο. 35 υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Δύο αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες, σταματάμε τις συνεδρίες μέχρι αύριο και ξεκινάμε αύριο στις 9. Καλό βράδυ.